Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η ψηφοφορία αύριο στις 11.30. Στην ημερήσια διάταξη τώρα έχουμε την έκθεση της κυρίας Φόρτ για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Να δώσω το λόγο στην συγγήτρια για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ σε όλους όσους συνεισέφεραν σε αυτή την έκθεση ε, και μέλη από διάφορες επιτροπές ε, και από περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανώσεις του κλάδου. Η εξέρεξη πετρελαίου αποτελεί ε, το 90% ε, του πετρελαίου και το 60% του φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι υψίστης της σημασίας για να μπορέσουμε να έχουμε ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια εφοδιασμού. Υπάρχει ε, μεγάλη ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές θάλασσες εκτός υδάτων και θα έπρεπε ε, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε εξορίξεις που θα μπορούσαν να έχουν ε, συνέπειες για τις θάλασσές μας. Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριλάβουμε και τις γείτονες χώρες ε, στα μέτρα που θα λάβουμε και η έκδοση αδειών θα πρέπει να είναι προτεραιότητα των κρατών μελών και όλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις οι οποίες είναι αντιφατικές και κάποια στοιχεία τα οποία είναι λανθασμένα. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τα διευκρινίσουμε αυτά πριν από την ψηφοφορία. Όλες οι πτυχές διαφέρουν. Δεν είναι επικίνδυνα απαραίτητα η εξόριξη ε, σε υπεράκτης δραστηριότητες και δεν είναι απαραίτητα ασφαλής η εξορίξη σε χαμηλά βάθη. Το ατύχημα του ε, Deep Waters και της BP μας έδειξε ότι υπάρχουν προβλήματα και θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα λαμβάνονται και όχι μόνο πριν από την οξέριξη αλλά για όλο τη, το κύκλο ζωής. Θα πρέπει να υπάρχουν επιθεωρήσεις και θα πρέπει να υπάρχει νομοθεσία που θα μας επιτρέπει να έχουμε συγκεκριμένους στόχους και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Το να ανταλλάσσονται ταχύτερα πληροφορίες μεταξύ ρυθμιστών και επιχειρήσεων είναι υψή τη σημασία, ιδιαίτερα για την πρόληψη ατυχημάτων. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένη νοοτροπία που θα επιτρέπει σε όλου να θέτουν ω προτεραιότητα την ασφάλεια και θα κάνουν κατάλληλο έλεγχο των ασφαλιστικών διαδικασιών και οι whistleblowers θα πρέπει να προστατεύονται. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε τι συνθήκες επικρατούν σε κάθε πλευρά. Ε, θα ε, πρέπει να υπάρχουν ρυθμιστές οι οποίοι να συναντώνται σε τακτά διαστήματα και θα πρέπει να υπάρχουν και πιο ε, καλά δίκτυα επιθεωρήσεων. Υπάρχει μια έκθεση η οποία όμως καταδεικνύει ότι αν έχουμε ένα νέο υπερρυθμιστή ε, πανευρωπαϊκά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε απαραίτητα καλά αποτελέσματα. Η καταστροφή του κόλπου του Μεξικού ε, και πολύ μεγάλο χρόνο καθαρισμού. Ε, πρόσφατα έχουμε βελτιώσει ε, ε, στον, εξοπλισμό καθαρισμού και κάλυψης και υπάρχει δυνατότητα να παρέχεται εξοπλισμός ε, καθαρισμού. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ταχύτατο εξοπλισμός αυτός. Ε, δυστυχώς η ΕΜΣΑ δεν έχει εμπειρία για πρόληψη ε, και προστατευτικό εξοπλισμό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ε, να διασφαλίσουμε ότι ο ρηπαίνων πληρώνει και οι επιχειρήσεις να είναι υπόλογες ε, και να αναλαμβάνουν το κόστος και τη ζημία, αλλά ορισμένες φορές θα πρέπει να υπάρχουν και δυνατότητα αμοιβαίων ασφαλιστικών ταμείων αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αγορά για να μπορέσουν να αγοράσουν εξωτερική ασφάλεια επιχειρήσεις. Η μελλοντική νομοθεσία λοιπόν όσον αφορά τις ε, οικονομικές ευθύνες δεν θα πρέπει να απαλλάσσει και, τους, ε, και τις μικρότερες επιχειρήσεις. Οι δυνατότητες για νέες εξορίξεις ε, και η απαγόρευση στην Αρκτική δεν είναι κατάλληλη. Θα πρέπει να, δούμε υπόψη, να έχουμε υπόψη και τι έγινε. Σε κάθε ε, περιοχή θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και θα πρέπει ε, να υπάρχει δυνατότητα εξόριξης όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι μπορούμε να διαχειριστούμε ενδεχόμενα προβλήματα. Αυτό ισχύει και για την Αρκτική αλλά και για οποιαδήποτε θαλάσσια περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μεστσάρος. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Φόρντ για την εξαιρετική έκθεση. Το Deepwater Horizon ήταν η καταστροφή της στην ανοιχτή θάλασσα που ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει πάλι τις λειτουργίες αυτές. Ο, η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τις ζημιές και εκείνη αναλαμβάνει το κόστος και όχι η κοινότητα. Η πρόληψη πρέπει να υπογραμμιστεί όπως και η αρχή της προφύλαξης η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη. Θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη καταστροφών και η ΕΜΣΑ θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για αυτές τις κέρυες λειτουργίες στην ανοιχτή θάλασσα περάκτης. Η συγκεντρωτική εποπτεία δεν σημαίνει ότι οι κανονισμοί θα εφαρμόζονται με τρόπο τέτοιο ούτως ώστε κάποιες εταιρείες να ωφελούνται ε, όταν είναι μεγάλες εν, ούτε θα πρέπει να υφίστανται διακριτικές ε, ε, αντιμετωπίσεις στις μικρές εταιρείες. Ευχαριστώ πολύ. domáce dodávky ropy a plynu majú významný prínos pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť a spotrebu energie v únii. viac ako 90 ropy a 60 plynu získavame práve prostredníctvom ťažby na mori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 Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρέπει να πω ότι οι παράκτιες γεωτρήσεις επηρεάζουν ενδεχομένως πολύ σημαντικά και άλλα κράτη-μέλη γειτονικά. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζονται κριτήρια απόδοσης πάνω σε θέματα ασφάλειας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να απολαμβάνουν υψηλού επίπεδου ασφάλειας και θα πρέπει να είναι απλοποιημένο το νομικό πλαίσιο λειτουργίας. Η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλύσουν λοιπόν τις πλέον προηγμένες πρακτικές σε θέματα ε, ε, άντλησης, ε, γεώτρησης και θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις. Ζητώ επίσης από τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν να διασφαλίζουν ότι τα καθεστώτα εξουσιοδότησης θα βλέπουν και την ύπαρξη ε, χρηματοδοτικών πόρων, ούτως ώστε να κινητοποιούνται πόροι εύκολα και γρήγορα για να αντιμετωπιστούν προβλήματα ε, στο περιβάλλον ή στην κοινότητα. Πριν δοθούν άδειε για υπεράντια γεώτρηση θα πρέπει να γίνουν μελέτες επιπτώσεων πάνω στο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φιγκερέιδο. Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε. Η εμπειρία που έχουμε και ο μεγάλος αριθμός ατυχημάτων δείχνουν ότι είναι επικίνδυνες οι υπεράκτιες γεωτρήσεις. Ο στόχος δεν είναι να αποκομίσουμε τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη από τις δραστηριότητες αυτές χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την ασφάλεια των εργαζομένων. Χρειάζονται λοιπόν σαφέστατοι κανόνες και για το περιβάλλον και βέβαια για τους ε, θυγόμενους εργαζομένους όπως και μέτρα προστασίας για τον πληθυσμό στην περιοχή αυτή. Αυτά πρέπει να είναι εγγυημένα. Είναι σημαντικό εδώ να έχουμε αποτελεσματική εποπτεία και να ακολουθούνται οι κανόνες κανονικά κάτω από ε, εντελεχή έλεγχο. Να μην λειτουργούν δηλαδή μόνο ε, για λόγους ιδιωτικού συμφέροντος ε, παραβιάζοντας το δημόσιο συμφέρον. Αυτό ε, πρέπει να το κάνει η Κομισιόν. Ο κύριος, η κυρία Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την κυρία Φόρντ για την έκθεσή της. Η ομάδα των Πρασίνων έχει ωστόσο καταθέσει εναλλακτικό ψήφισμα του οποίου ένα σημαντικό ε, τμήμα είναι η προστασία των ευαίσθητων περιφερειών και ιδίως τακτικής διότι αλλιώς θα είμαστε υπεύθυνοι διότι είδαμε τι συνέβη και στο κόλπο του Μεξικού βλέπουμε και στην Σκοτία τρομερές καταστροφές μέσα σε αυτά τα μοναδικά ε, θαλάσσια τοπία εξάλλου ποιος θα καθαρίσει τις περιοχές αυτές μετά από μια ενδεχόμενη καταστροφή αφού δεν πρόκειται για οικονομική ζώνη είναι ε, σε διεθνή ύδατα. Επισημένω ορισμένα προβλήματα. Τον έλεγχο πρώτα. Ασφαλώ και πρέπει να ενισχύσουμε τον έλεγχο. Ωστόσο, θα είναι καλό ο έλεγχο αυτό να είναι σε ευρωπαϊκή κλίμακα και να το αναλάβει ο Οργανισμό ε, Ναυτική Ασφάλεια. Δεύτερον, θέματα ευθύνη. Βλέποντα την τροπολογία 116, που την καταθέσαμε διότι προβλέπει πλήρη ευθύνη των ε, εταιριών πετρελαίου χωρίς οροφή. Έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν και οι περιβαλλοντικές ζημιές αλλά και οι οικονομικές και κοινωνικές ζημιές με υποχρεωτική ασφάλιση. Καλό είναι να σκεφτόμαστε τις μικρές πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά δεν έχουν ε, ασφάλιση, γιατί να τους δοθεί η άδεια εκμεταλλεύσεως. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά πράγματα και πρέπει να τα σκεφτείτε. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπο Σταγιάννη τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από το ατύχημα του Deepwater Horizon στον κόλπο του Μεξικού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο δράσεως για, να, για την προστασία και ασφάλεια του περιβάλλοντος σε περιοχές εξορίξεως πετρελαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε ευρέως τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση που συζητούμε σήμερα ε, επιβεβαιώνει την περιπλοκότητα του θέματος. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των δικών σας συμπερασμάτων και των συμπερασμάτων της Κομισιόν. Σας βεβαιώ ότι η Κομισιόν συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες σας σχετικά με την ανάγκη να αποφευθεί η αποσταθεροποίηση της ε, offshore εξόρυξης πετρελαίου με υπερβολική ρύθμιση. Πρέπει να διατηρηθούν οι επαφές με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξασφαλίζοντας έτσι ώστε οι προτάσεις μας να είναι και ρεαλιστικές και να άπτονται σε συγκεκριμένων σημείων. Η παραγωγή αερίου και πετρελαίου ε, σε υπεράκτιες περιοχές είναι σημαντική πηγή πλούτου και θα είναι για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και βεβαίω ε, έχουν και χαρακτήρα ιδιαίτερη υπεροχή οι ρυθμίσει ασφαλεία που διαθέτουμε. Θα συνεχιστούν οι προσπάθειε αυτέ. Η εμπειρία δείχνει ότι ποτέ δεν πρέπει κανεί να επαναπάβεται στι δάφνε του. Δυστυχώ η πρόσφατη διαφυγή ε, πετρελαίου σε έναν αγωγό τη Βόρεια θάλασσα, δείχνει ότι είναι ανάγκη ακόμα να ληφθούν δράσεις. Θεωρούμε ότι η ευθύνη των επιχειρήσεων πρέπει να μείνει στα χέρια του κλάδου και των εθνικών διοικήσεων. Η ανάλυση μας πάντως δείχνει ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε διάφορους τομείς πρέπει να εξασφαλίσουμε ώστε οι βέλτιστες πρακτικέ να επεκταθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενισχύσουμε την διαφάνεια του κλάδου και να προωθήσουμε την ανταλλαγή εμπειριών, να βελτιώσουμε τα σχέδια αντιμετώπισης επικουσών περιπτώσεων και προλήψεως. Αυτός μπορεί να είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως για να δώσει όθηση στην συνεργασία για τις βελτιώσεις αυτές. Ήδη έχει γίνει πολλή δουλειά με το σχέδιο πέντε σημείων για την ασφάλεια των υπεράκτιων ε, εξορίξεων που συνοδεύεται και από ανάλυση και μελέτη επιπτώσεων και θα υιοθετηθεί τον Οκτώβριο. Θα είναι στραμμένο στο μέλλον και θα επιτρέπει την ε, λήψη υπόψη των περιπλοκοτήτων του ισχύοντος συστήματος οι προσπάθειες αυτές πρέπει να υποστηριχθούν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρεται για τη θετική αντιμετώπιση του κλάδου. Διότι οι καταστροφές αυτές δεν γνωρίζουν σύνορα. Γι' αυτό και με τους διεθνείς εταίρους, κυρίως μέσα στο G20, εξακολουθούν οι προσπάθειες αυτές. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις προσπάθειές σας για την ενίσχυση της ασφάλειας στα ύδατα και θα συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις μελλοντικέ προτάσεις, οι οποίες όπως είπα θα κατευθούν τον Οκτώβριο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Αύριο στις 11.30 ψηφοφορία. Την ημερήσια διάταξη τώρα έχουμε την έκθεση της κυρίας Γιανακουδάκη για τις γυναίκες της ηθήνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια λοιπόν για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ.